Γιασένκο Σελιμόβιτς, Υγεία των Ζώων. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, κ. Σελιμόβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους και όλους ε, για την εξαιρετική αυτή δουλειά που έγινε. Το νομοθέτημα αυτό ήταν περίπλοκο, χρειαζόμασταν εμπειρογνωμοσύνη, ε, ήταν τεχνικό το κείμενο και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Επίσης να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Ήταν πολύ καλή, πολύ ευέλικτη στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια Επιτροπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφιέρωσε χρόνο και προσπάθεια. Καταφέραμε ένα εξασφαλίσουμε συμφωνία που ικανοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο νομοθετικό κείμενο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει στην πραγματικότητα για τη σχέση ανάμεσα στην υγεία των ζώων, την ανθρώπινη υγεία και την ε, ευζοία των ζώων. Οι μεταδοτικές ασθένειες, ε, ε, η γρήπη των πτηνών και άλλες μπορεί να επηρεάσουν και την για των ανθρώπων. Ε, το ίδιο και η αντιμικροβιακή αντίσταση. Η, η, η, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο γιατί θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε νόσους στο μέλλον. Μιλούμε επίσης και για τους γεωργούς. ο, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να ε, σέβονται τις αρχές ε, της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ε, τα κτηνιατρικά φάρμακα επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο λογικό, εύλογο και αναλογικό. Επίσης μιλάμε στο κείμενό μας για τα μέτρα που μπορούν να παίρνουν τα ε, κράτη-μέλη ε, προκειμένου να εμποδίσουν ε, την μετάδοση νόσων μέσω των αδέσποτων ζώων, σκύλων ιδίως, και να αποφεύγουν ταυτόχρονα βέβαια τις βλάβες επί των ζώων αυτών καθ' αυτών. Δίδεται επίσης η εντολή στην Κομισιόν ε, αν χρειαστεί στο μέλλον να δημιουργήσει ένα σύστημα, προτείνει ένα σύστημα καταγραφής των σκύλων. Επίσης ε, δίνουμε την, ε, στην Κομισιόν την δυνατότητα να παρέμει στην εφαρμογή μέσω κατεξοδότηση πράξεων. οι τεχνικές πτυχές ε, θα αφαιθούν στην Τεχνική Επιτροπή. Όλα αυτά είναι στο κείμενο που θα ψηφιστεί αύριο. Νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για να καταπολεμήσουμε το θέμα της, το πρόβλημα της ε, αντίστασης στα αντιβιωτικά. Ε, έχουμε πλέον ένα κείμενο με σαφείς στόχους που απλοποιεί την κοινοτική νομοθεσία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ε, κυρία Πόλσον εργάστηκε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Πόλσον. Ήταν η προκατοχός μου. Έχουμε μια συνένεση ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και ελπίζω το ίδιο θα συμβεί και αύριο στην Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Αντρουκάητης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου σήμερα με στόχο να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το έργο μας για τον κανονισμό για τις μεταδιδόμενες ζωνόσους που είναι ε, πιο γνωστή ως νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα στον τομέα αυτό, διότι έχει προκύψει μετά από πολύ σκληρή δουλειά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσμα είναι ε, από την κοινή προσπάθεια καταφέραμε να ε, κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η υγεία των ζώων και τι σχέση έχει με την ανθρώπινη υγεία. Επίσης αναγνωρίσαμε ότι οι επιδημίες ζωονόσων και κρίσεις μπορεί να συμβούν από καιρού καιρών. Επομένω, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό οτιδήποτε και αν μα επιφυλάσει το μέλλον και οποιασδήποτε ε, πιθανό σενάριο νόσου προκύψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη βιωσιμότητα του τομέα τη κτηνοτροφίας και τη υδατοκαλλιέργεια και επίση αυξάνει και την ανταγωνιστικότητά μα στι διεθνεί αγορέ. Η νέα νομοθεσία θα μας οδηγήσει σε ένα πιο αποτελεσματικό και εξορθολογισμένο σύστημα για την καταπολέμηση των ζωικών ε, την διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και επίσης ασφαλέστερη και πιο ε, ανταγωνιστική ε, δυνατότητα και περιβάλλον για τους γεωργούς μας. Επίσης θα υπάρχουν ευθύνε για όλους τους φορείς, για τους κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους και τις αρμόδιες αχέρ. Θα πρέπει να βελτιώνουμε την απάντηση στις επιδημίες ε, ζωικών νόσων και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλα μέτρα στον τομέα της ε, γεωργίας και της υδατοκαλοέργειας με αναλογικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή είναι καλά εγγεγραμμένη λοιπόν η βασική αρχή και αυτή τη στιγμή είναι όλο ένα και πιο βαθιά ριζωμένη σε σχέση για παράδειγμα με αυτά που κάνουμε για τη μικροβιακή εντοχή. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία αρχή για να εφαρμόσουμε τα όσα αποφασίσαμε για την υγεία των ζώων και τη στρατηγική 2007-2020. Δεν ήταν πάντα εύκολη διαδικασία, αλλά έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα και τα όσα περιλαμβάνουμε στο νέο πλαίσιο ε, τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά με όλου του ενδιαφορομένους και τα έχουμε εξετάσει ιδιαίτερα προσεκτικά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδε ε, και προσδοκίε για ευρεία συμφωνία στον τομέα αυτό. Σίγουρα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μα. θα υπάρξουν εκτελεστικέ πράξει και πράξει κατά εξουσιοδότηση, αλλά και η πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων αυτή τη στιγμή συμφωνηθούν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ε, είμαι ευγνώμων προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πολύ σημαντική συνεισφορά. Είναι σκληρή δουλειά και ε, μια επικοδομητική προσέγγιση από πλευρά Κοινοβουλίου μα βοήθησε να ε, φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτό το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συζητητέ, την κυρία Πόλσεν για την εξαιρετική επιτοχία τη ε, να καταφέρει επιτυχία σε πολιτικό επίπεδο, συμφωνία συγγνώμη, σε πολιτικό επίπεδο και επίσης ε, το γεγονός ότι συνεχίστηκε το έργο της κυρίας Πόλσεν και καταφέραμε να φτάσουμε το θέμα αυτό ε, στο τέλος του. Να ευχαριστώσω και τους σκιώδεις συγητές και από την προηγούμενη θητεία και από την παρούσα θητεία και την ομάδα των διαπραγματευτών για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν. Ελπίζω πλέον να μπορέσουμε να λάβουμε το τελικό βήμα και να εγκρίνουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα και να έχουμε ένα αίσιο πέρας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα θα μιλήσουν οι πολιτικές ομάδες. Εκ μέρους λοιπόν του ΕΛΚ, ο κύριος Ντες. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και τους και οδησηγητές ε, και σας τον Επίτροπο, κύριε Επίτροπε, όπως επίσης ε, και την προηγούμενη Προεδρία για την υποβολή αυτού του προγράμματος. Αυτός ο νέος κανονισμός για την υγεία των ζώων είναι προληπτική, είναι ένας ε, κανονισμός που συνδυάζει πολλές προληπτικές διατάξεις και θα οδηγήσει σε απλούστευση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Υπήρξαν πάρα πολλοί συμβιβασμοί, ε, συνοψίστηκαν και εξετάστηκαν πάρα πολλές ε, τροπολογίες και μπορέσαμε στην Επιτροπή Γεωργίας να επιτύχουμε μια ευρεία συνένεση όσον αφορά στην υγεία των ζώων. Είναι υποχρεωτικό Στη 28 κράτη-μέλη να γίνεται αναφορά θεμάτων που έχουν σχέση με την υγεία των ζώων, αλλά και ε, στη σχέση των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Για το δικό μας το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να ε, ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια για επιδημίες και για ασθένειες ζώων και αυτές οι διατάξεις να μεταφραστούν και να μεταφερθούν σε βασικό και θεμελιώδες δίκαιο. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι η επικαιροποίηση του καταλόγου των επιδημιών. Χαιρόμαστε που με αυτόν τον κανονισμό σίγουρα θα βελτιωθεί η δημόσια υγεία. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ευζοία των ζώων. Για τη δική μου την πολιτική ομάδα το σχέδιο αυτό ε, είναι άξιο του να το υπερψηφίσουμε και κύριε Επίτροπε είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη. Επόμενη η κυρία Τζουφρίντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με διάφορες ε, έκτακτες καταστάσεις, με επιδημίες που δείξαν ακόμα και σε θύμητα. Είχαμε την ε, επιδημία, την γρήπη των πτηνών, αλλά και πολλές άλλες ασθένειες ε, μεταδοτικές ασθένειες, νόση που αυτός ο κανονισμός έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναντέλφους που όπως και εγώ δούλεψαν πάνω σε αυτή την πρόταση. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Πόλσεν, ο οποίος με αυτόν τον κανονισμό κλείνει την εντολή του. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πραγματικά κατόρθωσε να επιτύχει μεγάλη συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δύο θέματα υπάρχουν που θέλω να υπογραμμίσω. Το πρώτο είναι ότι επιτέλους ε, τα πράγματα είναι ένα προμαύρο. Δηλαδή η υγεία των ζώων εξαρτάται από την ευζοία τους, από τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Ε, αν δεν υπάρχει καλή μεταχείρισή τους δεν θα υπάρχουν υγιή ζώα. Το άρθρο 13 της συνθήκης επισημαίνει ότι ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με κάποια λογική τα ζώα και όλοι αυτοί που τα αντιμετωπίζουν, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι άλλοι ε, θα πρέπει να νιώθουν ότι και αυτά υποφέρουν η ευζοία τους να είναι το πρώτο μέλημά τους ε, να ε, τα συμπεριφέρονται με ανθρωπιά. Κατόπιν, όσον αφορά τις μεταδοτικές νόσους, ε, η ζωοτεχνική η ζωτεχνία μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη, πρόληψη και μέσα από ιδιαίτερη υπευθυνότητα όσων ασχολούνται με τα ζώα. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός γιατί θα συσταθεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν, υπήρχαν κατά παρελθόν 40 νομοθετικές πράξεις, κάποιες μάλιστα ανάγονται και από την περιοχή της δεκαετίας, από την εποχή του 60. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τα ζώα και η υγεία τους και αυτό πόσο μάλλον σε μια Ευρώπη όπου έχουμε βασανιστήρια κατά των ζώων. Αυτά τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα πολύ συχνά και πολλοί μάλιστα τα ανέχονται ή κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Τζουφρίντα. Ο κύριος Βοχεχόφσκι παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και την κυρία Όλσον που δεν είναι παρούσα σήμερα πια. Η, το νομοθέτημα αυτό θα ασκήσει σημαντικότατη επίδραση στην υγεία των ζώων στην Ευρώπη και, ε, και στη δημόσια υγεία όμως, όχι μόνο στην υγεία των ζώων. Χαίρομαι εκ μέρους της ομάδας μου για το γεγονός ότι πολλές από τις ιδέες μας έγιναν αποδεκτές. Μιλήσαμε για τα δέσποτα ζώα, για τα κατοικίδια, για την υποχρέωση να καταγράφονται. Νομίζω ότι ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση το κείμενο. Βέβαια δεν είναι αρκετό Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Ε, ιδιαίτερα, για παράδειγμα, στην στήρωση των αδέσποτων ζώων που θα πρέπει να συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδοτείται. Ευχαριστώ. Ε, για τους φιλελεύθερους, ο Γιάνν Χουίτεμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Η αντιμικροβιακή ε, αντίσταση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το 70, 76% ε, ε, έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί η χρήση των αντιβιωτικών ε, στην κτηνοτροφία την τελευταία δεκαετία. Σε τέσσερα χρόνια όμως στην Ολλανδία μετά από τη λήψη μέτρων από την Ολλανδική κυβέρνηση σε τέσσερα χρόνια μειώθηκε κατά 15 περίπου Η υγεία των ζώων είναι συμφασμένη με την ανθρώπινη υγεία. Ε, αυτή την προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι προτάσεις των φιλελευθέρων νομίζω ότι βοήθησαν να υιοθετήσουμε σημαντικά νομιστικά κείμενα όπως ε, την ε, υπεύθυνη χρήση των αντιβιωτικών στην κοινοτροφία. Δεν είναι απλό. Χρειάζεται καινοτομία, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις από όλους. Δεν είναι δυνατόν ο ένας γεωργός να επενδύει και ο άλλος να μην επενδύει. η χώρα μου, οι κάτω χώρε είναι πρωταθλήτρια στη μείωση τη χρήση των αντιβιωτικών. Θα πρέπει να διδαχθούν οι άλλε χώρε από εμά. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Γκουε, τώρα ο λόγο του κύριο Στέφαν Εκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ομάδα τη Γκουε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή Αυτό που πρέπει να χαιρετήσουμε είναι ότι πρέπει να αποφεύγεται ο πόνος των ζώων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η δεσμευτική καταγραφή όλων των επαγγελματιών, κτηνοτρόφων ε, και των αγοραστών. Αυτό μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ε, το παράνομο εμπόριο των ζώων. Ε, γιατί υπάρχει αυτό το παράνομο εμπόριο με ζώα που δεν έχουν εμβολιαστεί ε, ζώα τα οποία δυστυχώς ε, οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται πάρα πολλούς κινδύνους και για την ε, διάδοση των επιδημιών. Πρέπει όμως δυστυχώς να πω ότι η πρόταση αυτή δεν εξυπηρετεί κατ' ουσίαν την προστασία των ζώων παρότι είναι σαφές ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην σωστή εμπορία και ε, στην σωστή διατροφή των ζώων. Περιμένουμε και προσδοκούμε από την Επιτροπή όταν μας υποβάλει ένα πλαίσιο το συντομότερο δυνατό δυνατόν για τη τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει ε, είναι ότι έχουμε εδώ ευαίσθητα όντα για τη δική μου λοιπόν την πολιτική ομάδα ε, είναι σημαντικό να οριστεί και το τι ακριβώς είναι αυτά τα ζώα για τα οποία συζητάμε ε, έχουμε τα δέσποτα ζώα αυτά αντιμετωπίζονται ως άγρια ζώα αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση της νομικής προστασίας των αδέσποτων ζώων και θα ήθελα πρώτα να σας υπενθυμίσω τι ακριβώς έχει γίνει στη Ρουμανία. Ευχαριστώ. thank you. On behalf of Greens, Deputy Bronis Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, naudodamasis progą noriu Jums padėkoti už atliekamą darbą šitoje srityje. Taipogi noriu padėkoti Τρέψατε μου επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση παρόλο που ε, το σχέδιο νομοθετήματος ε, ε, αποτελεί ένα μόνον πλαίσιο παρόλα αυτά αντανακλάω τις βασικές σκέψεις όσον αφορά την πρόληψη των επιδημιών. Υποστηρίζουμε ε, την ε, προστασία των ζώων όχι μόνο από νόσους αλλά και από πόνους και κακοποίηση. Ε, είναι σημαντικό ότι κατηγοροποιούνται διάφορες ασθένειες. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να λάβουν γνώση των διαφορετικών ε, προϋποθέσεων που μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την καλύτερη προστασία των ζώων. Αυτό που έχω κατά νου είναι τα έσοδα των ε, κτηνοτρόφων τα οποία συρρυκνώνονται συνέχεια για παράδειγμα όσον αφορά τους γαλακτοπαραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις στην υγεία των ζώων και ε, και σε ορισμένε ε, χώρες ε, μέλη οι γαλακτοφόρες αγελάδες δεν τρέφονται επαρκώς γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να τους παράσουν τα αναγκαία συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες κλπ. Και ε, βλέπουμε ότι οι οικονομικοί φάκτορες, ε, μπορούν να συμβάλλουν στην ε, διάδοση των επιδημιών. Άρα λοιπόν ε, θα ήθελα οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση και να, να αλλά θα πρέπει βεβαίως παράλληλα να βελτιωθούν οι οικονομικές προϋποθέσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ εκ μέρους ο Φιλίπ Λουασό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι η σύγχρονη επικαιρότητα μας έδειξε ότι η καλή διαβίωση των ζώων δεν τηρείται. Οι πρακτικές ορισμένων δεν ξέρουν ούτε να λάβουν υπόψη τα βασικά μέτρα. Θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα για την υγεία των ζώων και μέχρι το τέλος της αλυσίδας, διότι το διακύβευμα έχει να κάνει και με την ανθρώπινη υγεία, με την διατροφική αλυσίδα που απειλείται από την υγεία των ζώων. Το στρες, η κακή μεταχείριση, ο τρόπος φαγής ίσως αναπτύσσει επιδημίες όπως η κόλλη, η σαλμονέλα και αυτό εξαρτάται από τους ανθρώπους και από τον τρόπο που μεταχειρίζονται τα ζώα στην, ε, στην κτηνοτροφία, στον τρόπο μεταφοράς, στον τρόπο σφαγής. Οι κατοχώρες αποφάσισαν να έχουν αυστηρούς κανόνες για τα σφαγεία ε, και με ειδική σήμανση ε, διότι το να χρειάζεται πολλή, πολλή ώρα για να πεθάνουν τα ζώα είναι αντίθετο προς την καλή μεταχείριση των ζώων και τα μέτρα αυτά δεν τηρούνται από αυτές τις γερετολεστίες σφαγής. Έχουμε επίσης ορισμένα μικρόβια που προέρχονται από το στομάχι και από άλλα όργανα των ζώων. Θα πρέπει η Κομισιόν να λάβει μέτρα ούτω ώστε ορισμένε πρακτικές απαράδεκτες σε σφαγεία να μην είναι πλέον εφικτά αυτά τα μέτρα και αυτές οι συνήθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ντάτσα έχει τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον εισηγητή για την εργασία που έκανε για αυτόν τον σημαντικό θέμα, το περίπλοκο. Θα ήθελα να καλωσορίσω, να χαιρετήσω αυτήν την ε, έκθεση σχετικά που αφορά και τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες επιστημονικές αποδείξεις για την μικραβιακή αντοχή και το πώς να την αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι κτηνοτρόφοι να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις νόσους των ζώων. Είναι επιτακτική ανάγκη ε, να μην η αποτελεσματικότητα της παραγωγής να μην απειλείται ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της νομοθεσίας. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται εξίσου. Χρειάζονται ισότιμοι όροι και δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Εστέρ Γκαρσία. Αν Γκαρσία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή την εβδομάδα θα ψηφίσουμε σε δεύτερη ανάγνωση τη συμφωνία με το Συμβούλιο για την ζωική ε, για την υγεία μάλλον των ζώων και των φυτών, όπως είπε και η συνάδελφος Πόλσεν και όρισε κατά την προηγούμενη θητεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δράσει ε, πολύ αμεσότερα όταν ανακύψει μία ασθένεια. Υπάρχουν, υπάρχει ένας κατάλογος σημαντικών ασθενειών για να έχουμε καλύτερη νομική ασφάλεια οι κτηνίατροι θα διαδραματίσουν πιο σημαντικό ρόλο για την καταπολόμηση των ασθενειών και της ε, ε, ε, αντιβιωτικής αντοχής. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ασθένειες ανακύπτουν αλλά όσο πιο οργανωμένοι και προετοιμασμένοι είμαστε, για να τις αντιμετωπίσουν, τότε δεν θα μας πλήξουν τόσο. Δεν θα πλήξουν τα ζώα μας και εμάς, καθώς και την οικονομία μας. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και σε όλους όσους συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σάνι. Ναι, τη δέχεστε. Ο κύριος Σάνη έχει το λόγο. Ναι, κυρία Βουλευτά, αξιότιμοι συνάδελφοι, συμφωνώ ότι η παρούσα ρύθμιση εμφανίζει πολλά πλέον εκτήματα. Παρ' όλα αυτά έχω ένα ερώτημα. Μιλήσατε για την ευελιξία, αλλά σε ορισμένες χώρες υποστηρίζεται το σύστημα Τη προστασία των ζώων είναι αποκεντρωμένο, θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένο. Και αυτό καθιστά αδύνατη μια ενιαία στάση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε εδώ να υπάρχει ένας κίνδυνος. Έχετε τον λόγο. Αγαπητέ συνάδελφοι, προέρχομαι από μία από τις πιο αποκεντρωμένες περιοχές ε, της Ευρώπης στην Ισπανία. Άρα το θέμα δεν είναι η αποκέντρωση, αλλά ο συντονισμός και η οργάνωση. Αν η αλυσίδα λειτουργεί καλά, δεν ε, θα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει, εμείς διαθέτουμε ένα ευέλικτο σύστημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που ανακύπτουν άμεσα και πολλές φορές, όπως στην περίπτωση του E. coli, δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια άμεσα. Ε, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με την αποκέντρωση, υπάρχει πρόβλημα με την οργάνωση. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λανθασμένη χρήση αντιβιωτικών και η χρήση αυτών όχι για σκοπούς θεραπείας και ίασης δημιουργούν μικροοργανισμούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος από την ε, μικροβιακή αντοχή και αυτό το βλέπουμε στον ε, τομέα της πρόληψης και της ε, χρήσης εκ των προτέρων γιατί πολλές φορές ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κατά κόρον αντιβιωτικά. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ κρατών μελών έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε τα, τα σωστά στοιχεία στην Επιτροπή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να υπάρχει μείωση του κινδύνου από την αντίσταση στα μικρόβια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, μελέτες που να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Νίκολσον για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο κανονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα και να προστατεύσουμε την ζωική υγεία που έχει και επιπτώσει στο περιβάλλον. Στην δική μου περιφάρεια, την Βόρεια Ιρλανδία, έχουμε την οργάνωση η οποία θέλει να συζητήσει το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με την ζωική υγεία και επίσης το θέμα της ε, αντιμικροβιακής αντοχής. Επίσης όσον αφορά την φυματίωση των βοηδών στην ε, δική μου εκλογική ε, περιφέρεια είναι ένα σημαντικό ε, θέμα και δεν ξέρω τι γίνεται με την νομοθεσία στον τομέα αυτό. Υπάρχει όμως ένα θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο περιεκτικό ε, ολοκληρωμένο για το θέμα αυτό που θα εστιάζεται στην απλούστευση, στην ευελιξία, στην αντιμετώπιση της νόσου. Απλούστευση, εναρμόνιση της νομοθεσίας είναι καλό ε, παράδειγμα αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Ο εισηγητής επίσης από τη φοροτιμή στην Πόλσον ε, δεν είναι μεταξύ μας αλλά ήταν πάρα πολύ καλό μέλος ε, της Επιτροπής Γεωργίας και αυτό είναι φόρος τιμής των όσων έκανε για τόσο πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φράνσα Όμπερμαϊερ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω θα δείξετε την ίδια ανοχή αν ξεπεράσω και εγώ το χρόνο πριν, όπως ο προηγούμενος συνάδελφος. Ε, σύμφωνα με μια μελέτη ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση των ε, αντιβιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά θα πρέπει να συστήσουμε στους κτηνοτρόφους μια σύνεση όσον αφορά την χρήση των αντιβιωτικών. Το θέμα των αντιβιωτικών θα πρέπει να, γίνεται, να θίγεται και στο πλαίσιο των εμπορικών συμβάσεων. Σύμφωνα με ένα άρθρο της Νόη Τσούρχερ Zeitung, ε, στην Αμερική υπάρχει μια αύξηση της χρήσης των αντιβιωτικών. Ε, η προστασία της υγείας ε, προϋποθέτει μια ενιαία αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταναλωτές ε, δεν θέλουν να τρώνε κρέας το οποίο έχει μολυνθεί από την χρήση αντιβιωτικών. Ούτε μέσω της TTIP. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεώργιος Επιτίδιος. Η υγεία των ζώων είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με τον τρόπο που τα εκτρέφουμε όσο και με τον τρόπο με τον οποίο τα μεταχειριζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε να ελέγχουμε την ποιότητα των ζωοτροφών αλλά να εντοπίζουμε, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε νόσους οι οποίες μεταδίδονται σε αυτά και μετά μεταδίδονται στους καταναλωτές μέσω των ε, ε, προϊόντων που καταναλύσκουν κρέας, γάλα ε, και τυριά. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου αλλά και η κλιματική αλλαγή εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για την υγεία των καταναλωτών. Και γι' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απλοποιήσει, ε, να ε, εντατικοποιήσει τους ελέγχους στα ζώα τα οποία εισάγονται από χώρες που δεν ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά παράλληλα να μην μεταδίδονται και οι νόσοι στους καταναλωτές για την αναγκαιότητα αυτού του πράγματος θα να αναφέρω ως παράδειγμα την χώρα μου την ελλάδα στην οποία εισάγονται πολλές φορές λαθρέα ε, εγωπρόβατα κυρίως από την τουρκία αλλά και από τα σκόπια τα οποία δεν έχουν υποστεί τους προβλεπόμενους ελέγχους άρα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εγχωρίων φυλών των ζώων αλλά και των καταναλωτών. αντιθέτως αυτά που εξάγονται από την ελλάδα είναι εγγυημένα. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μαριάννα Πετήρ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτήν την έκθεση. Η υγεία των ζώων είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχούμε λόγω ε, της αύξησης της ε, μικροβιακής αντοχής. Είναι μεγάλη απειλή για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Και έχουμε νέα στελέχη βακτηριδίων ε, που αντέχουν στα, μικρο, στα, στα φάρμακα, που αντέχουν στα αντιβιωτικά και επίσης οι καταναλωτές εξαρτώνται από την τροφή που καταναλύσκουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερήφανη για τα πρότυπα που υπάρχουν. Έχουμε διάφορες συμφωνίες παγκοσμίου εμπορίου και ε, μια ρύθμιση είναι αντίδραση στην υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών θα πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία ε, συγκριτικά σχετικά με την χρήση των αντιβιωτικών στα κράτη-μέλη. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μειώσουμε την αντιμικροβιακή αντοχή. Οι εκτινοτρόφοι θα πρέπει να ε, διατηρήσουν τις καλές κτηνοτροφικές ε, ε, πρακτικές. Έχουμε λοιπόν και εδώ ε, την διάσταση της ανθρώπινης υγείας. Εκτός από την υγεία των ζώων έχουμε ε, συνέπειες πάνω σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Μια μπλε κάρτα. Την δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ναι. Από τον κύριο Λεμπρετό. Ο κύριος Λεμπρετό έχει τον λόγο. Δέχεστε την ερώτησή μου. Κυρία Πετήρ, Τονίζεται ότι είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε την μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών, αλλά δεν είναι η αγροτική πολιτική της Ένωσης που ενισχύει και ενθαρρύνει αυτήν την χρήση. Έχει δημιουργήσει βιομηχανίες, μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες όπου περιορίζονται τα ζώα. Αυξάνεται έτσι η κατανάλωση των αντιβιωτικών και αυξάνεται η απειλή ε, για την ανθρώπινη υγεία. Δεν είναι ένα άλοθη αυτό ε, για να αποκρύψουμε την μεγάλη αποτυχία της αγροτικής πολιτικής της Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι η ΚΑΠ είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, οι αγρότες μας χρησιμοποιούν αντιβιωτικά ε, κατά διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια τροφίμων, η διατροφική ασφάλεια και είμαστε περήφανοι για την διατροφική μας ασφάλεια. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά επίπεδα θα πρέπει να γίνει συνετή χρήση αντιβιωτικών. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι δύο χρόνια μετά την πρώτη ανάγνωση φτάνουμε σε μία συζήτηση και τελική έγκραση του κανονισμού. Ο κανονισμός είναι ύψης της σημασίας μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ γιατί αναφέρεται στην υγεία των ζώων και φυσικά και στο ζωικό μας κεφάλαιο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές μας. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Πόλσεν που ε, δεν είναι μαζί μας και τον κύριο Σελιμόβιτς για την επιτυχία αυτού του κανονισμού. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ε, ε, αντιμικροβιακή αντοχή και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς χειριζόμαστε και τις ζωοτροφές, ιδιαίτερα τις ζωοτροφές που εμπεριέχουν φάρμακα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες και να υπάρχει ιχνηλασιμότητα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κοράτσα Πίλτ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστηρίζω πλήρως αυτό το νέο νομοθέτημα γιατί ε, ε, η αντοχή στα αντιβιωτικά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Πολλοί καταναλωτές ανησυχούν για το γεγονός ότι ε, στα ζώα χρησιμοποιούνται πάρα πολλά φάρμακα και είναι πολύ σημαντικό που το θέμα αυτό συνδέεται τώρα με την ανθρώπινη υγεία και με τον τρόπο τρόπο αυτό μπορούμε επίσης να αποτρέψουμε τις ε, ζώνες ούτως ώστε να μην σφαγιάζονται άρρωστα ζώα. Θα πρέπει να προσθεθούν κατά την άποψή μου τα... οι κανόνες και θα πρέπει ή δυνατόν να χρησιμοποιούνται, ε, ή δυνατόν να περιοριστεί η χρήση των αντιβιωτικών. Και είναι πολύ ε, σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε ποια ακριβώς φάρμακα χορηγούνται ούτε ώστε να διευκολύνεται και ο ανταγωνισμός. Ε, κάρτα από την κυρία Ντέσ, από την ίδια πολιτική ομάδα. Ναι, ε, κυρία συνάδελφε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε μαζί μου στο εξής. Στην κτηνιατρική έχουμε, μια πολύ, έχουμε ένα πολύ αυστηρό κανόνα τεκμηρίωσης. Ε, ίσως ε, θα έπρεπε οι αυστηροί αυτοί οι κανόνες να διευρυνθούν και στην ανθρώπινη ιατρική γιατί είναι πολύ σημαντική και η προστασία της υγείας των ανθρώπων. Συμφωνείτε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέσσε. Ναι, όπως σας είπα, ε, πολύ πραγματικά ανησυχούν για την ε, υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών τόσο στα ζώα όσο και στα ανθρώπινα όντα και ε, βεβαίως ο κανονισμός αυτός αφορά τα ζώα αλλά εδώ γίνεται μια ξεκάθαρη διασύνδεση με την ανθρώπινη υγεία και βασίζεται και στην επιστήμη ότι μπορούν, ε, μπορούν οι κίνδυνοι να μεταφερθούν από τα ζώα στον άνθρωπο. Ε, γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο σημαντική αυτή η νομοθεσία. κύριος Σεράου Σάντος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στην πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών στα ζώα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αντιμικροβιακή αντοχή ιδιαίτερα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δε μεταδίδονται αυτά αυτές και στον άνθρωπο μέσα στα πλαίσια της αντιμικροβιακής αντοχής όπως ε, ε, ε, μας ενημέρωσε το περιοδικό, το έγκριτο περιοδικό The Lancet με βάση μία μελέτη που διενεργήθηκε στην Κίνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να δούμε κατά πόσο διαβιβάζονται και μεταβιβάζονται ασθένειες ε, εξαιτίας του γεγονότος ε, ότι υπάρχει μεγάλη αντοχή στα μικρόβια από την υπερβολική χρήση των ε, αντιβιωτικών. Πρέναν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο νόμος, ο κανονισμός που θα ψηφίσουμε αύριο σχετίζεται με δύο ανησυχίες που έχουν εκφράσει και οι ψηφοφόροι μας. Μας ενδιαφέρει η ε, προώθηση της υγείας των ζώων και φυσικά να αντιμετωπίσουμε και τα αδέσποτα. Ως προς τις ασθένειες των ζώων ε, δεν υπάρχει κάποια διάρθρωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύει περισσότερο ή λιγότερο το Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για να έχουμε κοινού κανόνες σε περίπτωση εκδήλωσης ασθενειών. Επίσης, ως προς τα αδέσποτα, θα πρέπει να υπάρξει ανάθεση ευθυνών από τις, αρχικές, από τις εθνικές αρχές καθώς και ανθρώπινη αντιμετώπιση των δέσποτων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και το θέμα της υγείας αλλά και της ευζοίας των ζώων. Κάτι το οποίο ισχύει και για τα ζώα όπως ισχύει και για τους ανθρώπους. Μπαίνουμε στη διαδικασία catch Α, μπλε κάρτα, μπλε κάρτα. Δέχεστε ε, μία μπλε κάρτα από την κυρία Γκραπίνη. Από την κυρία Γκραπίνη. Δέχεστε μπλε κάρτα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας υποβάλω μία ερώτηση γιατί ε, χαίρομαι που θέσατε το θέμα των αδέσποτων, ιδιαίτερα των σκυλιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας μας έχει τη δική του εμπειρία. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το θέμα της υγείας των αδέσποτων. Έχετε κάποιο τρόπο να μας προωθήσετε, διότι το ζήτημα είναι ε, το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα των αδέσποτων γενικότερα. Μπράνεν. πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Τα σκυλιά δεν γνωρίζουν το χώρο Σέγγεν και θα μπορούσαν να διαβούν τα σύνορα τη στιγμή που δεν υπάρχουν εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εάν οι χώρες μεμονωμένα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αδέσποτων δεν θα τα καταφέρουν. Μόνο με συνεργασία μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε και τις συναφήνες ασθένειες. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλεμπαχ για ένα λεπτό. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Έστω και αν ε, στην προηγούμενη συζήτηση ορισμένοι συνάδελφοι αρνήθηκαν ότι η πολιτική υγεία είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση, ωστόσο αυτή η συζήτηση έδειξε πολύ καθαρά ότι η πολιτική υγεία ε, σαφώ είναι μια κοινή ε, πολιτική και κοινή ευθύνη των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην πολιτική υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσει μεταξύ των χωρών μελών. Θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση των ζώων και των ανθρώπων και αυτό το πακέτο οδηγεί στην αποφυγή της μετάδοσης των νόσων και δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούμε μόνο μέσω της συνεργασίας να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Η υγεία των ζώων προϋποθέτει ε, να έχουμε καλές ε, πρακτικές ε, εκτροφής των ζώων που γίνεται αντικείμενο ελέγχων και εποπτείες. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων, των κτηνικών φαρμάκων στα ζώα. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα ε, διακινούνται δια της Ευρωπαϊκής, ε, μεταδίδονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γνωρίζουν όρια. Και ένα ερώτημα και υποθέτουμε λοιπόν ότι μια αποτελεσματική προστασία των ζώων θα οδηγήσει σε μια καλή υγεία ζώων και ανθρώπων. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Σε υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει αρχικά να αυξηθούν τα μέτρα πρόληψης και μείωσης των επιπτώσεων των ασθενειών των ζώων. Θα πρέπει δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να προωθήσουν πρακτικές κτηνοτροφίας και καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να μειωθούν τυχόν απειλές για τη δημόσια υγεία επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα διάφορα είδη επιτήρηση που διενεργούν οι ομάδε που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη υγεία των ζώων ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Τέλο θα πρέπει να υπάρξει ένα απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο στην ευρωπαϊκή ένωση για την προστασία τη υγεία των ζώων τη δημόσια υγεία, αλλά και τη καλή διαβίωση των ζώων και αυτό σημαίνει πέραν των άλλων μείωση τη χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία χρήση κατάλληλων ζωοτροφών και έλεγχο της εισαγωγής ζώων και κυρίως προβάτων από την τουρκία και τα σκόπια όπου η νόση των ζώων είναι διαδεδομένη και όπου δεν υπάρχουν επαρκείς υγειονομικοί έλεγχοι των ζώων. μάλιστα αρρώστιες προβάτων από την τουρκία έχουν μεταδοθεί στον εύρο και σε άλλες περιοχές της ελλάδας με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιά οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο έλληνες κτηνοτρόφοι οι οποίοι θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν και να τύχουν της οικονομικής στήριξης της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ε, gospodine predsjedavajući dugi popis bolesti životinja Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο ασθενειών των ζώων που πλήττουν την ευημερία τους και να πλήξουν και την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, η γρήπη των πτηνών, η πανόλης των χείρων που πλήττει και ανθρώπους. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός είναι πολύ καλός διότι ορίζει μία καλή ισορροπία μεταξύ ευημερίας των ζώων και ανθρώπινης υγείας. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανθρώπινης ε, υγείας μαζί με την υγεία των ζώων. Γι' αυτό ελπίζω η Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πανευρωπαϊκά. Ε, Τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα των ανθρώπων, τότε αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος ε, μετάδοσης νόσων από τα ζώα. Αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση της Αφρικανικής Πανόλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει τα κονδύλια κατά 10% για την αντιμετώπιση αυτών των νόσων. Τα καλά λόγια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά εμείς λέμε ότι ε, ο, διάβολος έχει πολλά πόδια. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει διατροφική ασφάλεια και αυτό θα πρέπει να το δούμε και με στα πλαίσια του TTIP γιατί διαφορετικά η συζήτηση αυτή δεν θα είναι παρά μία κενή πρωτοβουλία που δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Ομπάμα μίλησε για αυτήν την αντιμικροβιακή αντοχή ε, και την έθεσε ως προτεραιότητα. Ε, θα πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε για το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό το θέμα αυτό είναι ε, σχετικά με την κτηνοτροφία και την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Αυτό που ως το 2050 ε, ατελείωτη τόνοι αντιβιωτικών θα χρησιμοποιηθούν για τα ζώα, 40.000 κατέτος. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα αυτό έχει σχέση με τα δικαιώματα των ζώων, τα δικαιώματα των ανθρώπων και τα δικαιώματα όλων μας. Πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών που επηρεάζονται από αυτήν την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών. Ευχαριστώ. Πίρκο Ρούχολεν Ρέρνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό για την υγεία των ζώων ενέχει ιδιαίτερη σημασία διότι για πρώτη φορά υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ζωική υγεία και στην ανθρώπινη υγεία. Στρεφόμαστε προς το μέλλον. Υπάρχουν νόσοι που μεταδίδονται από ζώο σε ζώο ή από ζώο σε άνθρωπο. Και αυτή είναι η απειλή του 21ου αιώνα. Η εργασία του κυρίου Σελίμοβιτς είναι πάρα πολύ καλή. Έχει προτάξει το γεγονός ότι χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα στην χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Τα αντιβιωτικά είναι επικίνδυνα. Πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα αντιβιωτικά και γνωρίζουμε όλο και περισσότερα πράγματα κάθε μέρα και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος Ήταν ο τελευταίος ομιλητής και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επίτροπης ο Επίτρος Άντριου Ακάτης. Κάιτης. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πάουλσολ και τον κύριο Σελίμοβιτς, ε, τους κοιόδης εισηγητές για την εξαίρετη εργασία. Άκουσα ε, ε, τη συζήτηση με πολύ προσοχή, τα διάφορα επιχειρήματα, τα διάφορα σημεία και είδα την ενδιαφέρον που επέδειξαν τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφερθήκατε στην οικονομική κατάσταση. Η Επιτροπή γνωρίζει ποια είναι η οικονομική κατάσταση που ε, σε ορισμένες ε, ε, περιπτώσεις έχει επίπτωση στην ζωική υγεία. Έχουμε το θέμα των αδέσποτων ζώων και θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες με ταυτοποίηση των ζώων αυτών, των αδέσποτων και άλλα ζώα που είναι και οικιακά ζώα. Νομίζω ότι έχουμε το νομικό πλαίσιο με τον νέο νόμο που περιλαμβάνει βασικούς κανόνες για την ταυτοποίηση, την καταγραφή των ζώων και για τα είδη των ζώων όπου τα, οι κανόνες ταυτοποίησης και καταγραφής υπάρχουν τώρα, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρξουν περαιτέρω απαιτήσει λεπτομερείς για την ταυτοποίηση, τα γραφή ζώων, άλλων ειδών, ε, σκύλων, ε, ε, για, για τα οποία δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσει τώρα. Η αναγκαιότητα θα εκτιμηθεί από την Κομισιό ε, μετά την υιοθέτηση του νόμου για την ζωική υγεία. Έχουμε δεσμευθεί για την καλή μεταχείριση των ζώων. Είναι το θέμα πάρα πολύ σημαντικό όπως το αναφέρατε στη συζήτηση. Βεβαίως εστιάζεται εδώ στις μεταδιδόμενες ασθένειες, μεταδοτικές ε, και δεν ρυθμίζει ακριβώς ε, την καλή διαβίωση των ζώων. Θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις διαμέσου ε, τριμερούς ε, διαλόγου για να ε, αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου για την καλή μεταχείριση των δόντων. Δεν ήταν πάρα εύκολο να συμφωνήσουμε για όλα τα σημεία, αλλά κατανοούμε την σημασία που έχει το θέμα αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάναμε μια ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Έχουμε καλύπτουμε διάφορα είδη, διάφορα της, της οτόκες, όρνηθες, ο παραγωγής κοτόπουλα, κρεατοπαραγωγής και άλλα. Αμερικοί στην, αναφέρθηκαν στην μικροβιακή αντοχή που είναι σημαντική για μένα τα θέμα αυτό θα περιλαμβάνεται πάντοτε στην πρόταση της Κομισιόν για την υγεία των ζώων ε, και για όλα τα φάρμακα, ούτω ώστε θα έχουμε μια καλή βάση για το θέμα αυτό. Επίσης η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση. Η Κομισιόν αναλαμβάνει ε, να εκδίδει μια τακτική έκθεση σχετικά με την χρησιμοποίηση αντιμικροβιακών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των στατιστικών των κρατών μελών και βεβαίως θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει συμφωνία δεύτερης ανάγνωσης για το θέμα αυτό που θα διανοίξει τον δρόμο για τα πολλαπλά πλέον εκτήματα που θα προκύψουν το σύντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα νομίζω θα δώσουμε τον λόγο ε, στον εισηγητή τον κύριο Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, υποστήριξή σας και θα ήθελα να τονίσω και πάλι πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια συμφωνία γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τη βαθμό συμφωνία σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημιουργείται και μια διασύνδεση μεταξύ υγεία των ζώων και δημόσια υγεία. Και μελλοντικά με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο στα χέρια μας για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις ε, επιδημίες των ζώων. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους για την υγεία τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων και με τον τρόπο αυτό επίσης μπορούμε να εξοικονομήσουμε και πολλά χρήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλους σκοπούς. Εάν υπερψηφιστεί η έκθεση, αυτό είναι σημαντικό βήμα όσον αφορά την καταπολέμηση της μικροβιακής ε, της αντοχής και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είναι θετικό ότι πάρα πολλές ε, οργανώσεις ε, υποστηρίζουν η ΚΟΖΕΚΑ, ε, πολλοί σύλλογοι νόσης προστασίας των ζώων, κτηνιατρικές ενώσεις κλπ. Και αυτό αποδεικνύει ακριβώς πόσο σημαντική ήταν αυτή η συμφωνία και ελπίζω το Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτό το νομοθέτημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τους όδης, τον κύριο Επίτροπο και όλους όσους ε, συνέβαλαν θετικά σε αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ.